διάταξης ε, δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την Κούβα. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον ε, Υπουργό τον εκπρόσωπο τη Επιτροπή ε, και να πάμε στην επόμενη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον Υπουργό για τη δήλωσή του. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο θάνατος του Ορλάντο Θαπάτα υπήρξε ένα ε, ιδιαίτερα αρνητικό γεγονός. Ένα γεγονός που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί και δεν θέλουμε να ε, ξανασυμβεί ε, όχι μόνο στην Κούβα αλλά σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Ο, η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών είναι ακριβώς να καταγγείλουμε τα γεγονότα αυτά που αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εργαστούμε έτσι ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το γεγονός ποτέ. Αυτή πρέπει να είναι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, ως βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό, ε, γιατί πιστεύουμε στις αξίες της ελευθερίας, της ε, ανοχής, του πλουραλισμού και ε, γι' αυτό ε, αυτά αποτελούν έκφραση της, γνήσια έκφραση της προσωπικότητάς μας. Εκεί λοιπόν όπου, προκύπτουν αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι καθολικά, το, το καταγγέλουμε, το καταγγέλουμε φωναχτά και αυτό το κάναμε και όσον αφορά την Κούβα όπου εκφράσαμε την απεσιοδοξία μας και την βαθιά μας ανησυχία για την έλλειψη προόδου στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Το είπαμε επίσης όταν απαιτήσαμε την απελευθέρωση των ε, ε, πολιτικών κρατούμενων στις φυλακές της Κούβας. Γύρω στους 200 ε, τέτοιους φυλακισμένους έχει η Κούβα αυτή τη στιγμή. Ορισμένοι, ορισμένοι η κατάσταση υγείας είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται σε απεργία πείνας. Αυτό το, το κάναμε όταν τονίσαμε ε, ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Το πράξαμε όταν ε, μιλήσαμε για το θάνατο του Ορλάντο Θαπάτα και είπαμε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο ε, αφορά την ίδια την ευθύνη μια κυβέρνηση που έχει τέτοιου κρατούμενου. Πάντω η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Κούβα είναι κάτι περισσότερο. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διαρθρώνεται γύρω από συγκεκριμένα στοιχεία και εγώ ε, θα ήθελα να τονίσω ορισμένα από αυτά. Πρώτα απ' όλα, ο πολιτικός διάλογος. Ε, πολιτικός διάλογος με τους θεσμούς της Κούβα, με τις αρχές και με το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών γιατί και αυτά βεβαίω τα θέματα ε, συμπεριλαμβάνουν, του διαλόγου συμπεριλαμβάνουν και, τον, ε, ε, και, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, η, η αναπτυξιακή συνεργασία, που είναι αλληλεγγύη προ τον κουβανικό λαό. Και τέλο, να προωθήσουμε τι αλλαγέ στην οτροπία και στη δημοκρατική πρακτική στην Κούβα. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα στοιχεία τη πολιτική μα, μια πολιτική που που έχει ένα βασικό αποδέκτη, τον λαό της Κούβας, ε, με στόχο την ευημερία του, την πρόοδο, ε, την ε, βελτίωση των συνδικών διαβίωσης και κυρίως την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η Επίτροπη λυπάται για τον θάνατο του Ορλάντο Ζαπάτα και τις περιστάσεις αυτού του θανάτου και θα ήθελα να εκφράσω επίσης την ανησυχία μου για τους άλλους πολιτικούς κρατούμενους στην Κούβα. Όλοι εδώ ε, συμμεριζόμαστε ε, το ίδιο συνέστημα απογοήτευσης ε, και οργής μετά το θάνατο του Ορλάντο Ζαπάτα και δεν θα πρέπει να αφιστούμε καμιά προσπάθεια ούτω ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό στην Κούβα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις αξίες της δημοκρατίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών που προσπαθούμε να προτεστατεύσουμε και να προωθήσουμε αφού υποφέραμε από παραβιάσεις αθεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολύ πρόσφατα στην Ήπειρό μα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια και δεν έχουν σύνορα. Αυτή η αρχή είναι αναπόσπαστο μέρος του διαλόγου μας με όλους τους εταίρους στην Ευρώπη και εκτός της Ευρώπης η επικοδομητική ε, δέσμευση, όχι μια πολιτική καταπίεση και κυρώσεων, αποτελεί τη βάση της ε, πολιτική μας απέναντι στην Κούβα, όπω τονίστηκε ε, στην κοινή θέση που υιοθετήθηκε το 1996. Αυτό είναι η λογική που σύμφωνα με την οποία αποφάσισε η Κομισιόν Άρη το 2009 τα, τις κυρώσεις του 1993 ούτως ώστε να διευκολύνει το διάλογο και να επιτρέψει την πλήρη χρήση των μέσων της κοινή θέση του 1996. Επίσης, πάρα πολλά κράτη-μέλη μπορούν να συνεχίσουν ε, την αναπτυξιακή συνεργασία με την Κούβα ε, τα τελευταία ε, μήνες και αυτό αντανακλά την κοινή άποψη για την σημασία που πρέπει να παίξει η αναπτυξιακή συνεργασία με την Κούβα. θα ήταν η χειρότερη λύση για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το σταματήσουμε αυτό. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η αξιοπιστία μας ως παίκτη, αλλά και η ικανότητά μας να είμαστε παρόντες στην Κούβα. Πιστεύω ακράδαντα ότι για να προχωρήσουμε θα πρέπει να εμβαθύνουμε στον πολιτικό διάλογο και στην συνεχιζόμενη συνεργασία με την Κούβα ως εργαλείο για να βελτιώσουμε τη ζωέσα του κουβανικού, των κουβανών πολιτών. Η συνεργασία ποτέ δεν διακόπηκε με την Κούβα. Γιατί, διότι η ανάπτυξη δεν είναι υποστήριξη στην κυβέρνηση, είναι υποστήριξη στο λαό. Η άποψή μας ήταν πάντοτε ότι η αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί σημαντικό στοιχείο των σχέσεών μας με την Κούβα το συνεχιζόμενο σχέδιο με την Κούβα ωφελεί άμεσα στους πληθυσμούς καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες με την υποστήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον κυκλώνα με την διατροφική ασφάλεια και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επίσης υπάρχουν έργα και προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν δραστηριότητες από μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Δεν υπάρχει ε, δεν υπάρχει χρηματοδότηση σε δημόσιες αρχές ε, δίνονται τα χρήματα σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικέ οργανώσεις και σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που χαιρετίζουν την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κούβα. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθήσει να ασχολείται με τις βασικές ανάγκες του κουβανικού πληθυσμού ε, με παρέμβαση σε στρατηγικούς τομείς με διάφορα μέσα γεωγραφικά και όλα. Το να προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα μέσα στον διάλογο, υποστήριξη ε, του λαού διαμέσου της ε, συνεργασίας αναπτυξιακής ε, και και η παρουσίαση των αρχών μας είναι ο τρόπος. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Σαλαφράγκα για την ομάδα του ΕΛ και δυόμιση λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, όταν η πολιτική, μου, η πολιτική ομάδα ζήτησε την συμπερίληψη θέματο στην ημερήσια διάταξη, δεν το πράξαμε για να ε, τονίσουμε ε, τα ανεπανόρθωτα σφάλματα μερικέ φορέ των πολιτικών ε, που είναι συγκαταβατικέ απέναντι στου εχθρού τη ελευθερία. Ούτε θέλαμε να αποκομίσουμε πολιτικά ωφέλη. Το πράξαμε διότι το κοινοβούλιο μα, που είναι ο θεσμό, η η ύψιστη έκφραση τη δημοκρατία στην Ευρώπη, να καταδικάσει το θάνατο ενό αθώου και κυρίω να εκφράσει την αλληλεγγύη του απέναντι σε όσου στην Κούβα αγωνίζονται, ζουν και, ε, ε, και πεθαίνουν, όπω ο Ορλάντο Θαπάτα, για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του. Όπω υπενθύμησε και πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, υπάρχει, έχουμε την κοινή θέση του Συμβουλίου που είναι αξιοσέβαστη, διότι ζητεί την άμεση και χωρί όρου απελευθέρωση των πολιτικών κρατούμενων και συνεκτική, διότι ζητά να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα και θεμελιώδει ελευθερίε έτσι ώστε ε, να προσελκύσουμε την Κούβα στο δικό μας το σύστημα αξιών και όχι σε συστήματα άλλων όπως η Κίνα. Ε, όμως εδώ αντιχούν τα λόγια ενός ε, γενναίου ε, ανθρώπου ε, του ε, βραβευθέντα με το βραβείο Ζαχάροφ το 2001. Η πρώτη, ο πρώτος θρίαμβος της ελευθερίας είναι να μην υπάρχει μίσος στην καρδιά των ανθρώπων. Να μην, να μην μισούμε τους συνανθρώπους μας. Σε αυτό αναφερόταν. Και ο Αντρέη Ζαχάροφ άφησε κλειοδότημα ελευθερίας και υπέρ, υπέρ της ελευθερίας των λαών. Και μερικές φορές οι φωνές, οι πιο σημαντικές είναι οι φωνέ που δεν ακούγονται. Εδώ δεν μπορέσαμε να ακούσουμε τι φωνέ ε, των Δάμπα Δεμπλάνκο που επίση ε, πήραν το βραβείο Σαχάροφ. Ε, δεν, μπορούσαμε, δεν μπορέσαμε να ακούσουμε ούτε και τη φωνή του Ορλάντο Θαπάτα. Αλλά σύντομα θα μπορέσουμε να ακούσουμε τη φωνή πολλών άλλων κουβανών. Στο μεταξύ, κυρία Πρόεδρε, το κοινοβούλιο μα με την νομιμότητα που έχει διότι εκπροσωπεί 500 εκατομμύρια πολιτών από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ε, εκφράσει σαφώς ε, αυτή την κραυγή ελευθερίας που έρχεται, που έρχεται από το αγαπημένο νησί της Κούβας. Σας ευχαριστώ. Thank you. On of the... Ευχαριστώ. Τώρα, ο κύριος Γιάννης Μπαρνουέβο Γκάρση, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε του Συμβουλίου, Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, να μην επιτρέψουμε ποτέ η σιωπή μας να μετατραπεί σε ε, συνενοχή ε, με αυτούς που σκοτώνουν την ελευθερία ποτέ πια ένα ένας άνθρωπος που αγωνιζόταν για τα δικαιώματά του και τα δικαιώματα των υπολείπων να μην πεθάνει στις φυλακές της Κούβας ή το οπουδήποτε αλλού χωρίς να, να υψώσουμε τη φωνή μας με αποφασιστικό τρόπο και να απαιτήσουμε ε, την ε, διάσωση των ανθρώπων αυτών. Ο κύριος Ορλάντο Θαπάτο, ένας ε, πολίτης 42 ε, ετών που το μόνο που ζητούσε ήταν να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης μετά από 86 μέρες απεργίας πείνας και 7 χρόνια φυλακής πέθανε ακριβώς γιατί ζητούσε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σε αυτά τα 7 χρόνια υπέστη κακομεταχείριση, ε, ταπείνωση ε, από τους ε, δεσμότες του μέσα σε βαριά σιωπή από τη διεθνή κοινότητα. Άλλοι ε, αγωνιστέ στην Κούβα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση απεργία πείνα, όπω ο, ο Γκυγέρμο Φαρίνια, δημοσιογράφο και ψυχολόγο. Κυρίε και κύριοι, το ψήφισμα το οποίο υποβάλλουμε σήμερα ε, και το οποίο ε, θα υποβάλλουμε σήμερα θα ψηφίσουμε αύριο και το παρουσιάζω εγώ εξ ονόματο τη ομάδα των Σοσιαλιστών, ζητά την απελευθέρωση όλων των, ε, των, των κρατούμενων συνείδηση στην Κούβα. Επίση να υπάρξει άμεση μετάβαση προ τη δημοκρατία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή δεν υπησερχόμαστε σε ένα, σώμα, σε ένα θέμα που μα διαιρεί το κατά πόσο θα πρέπει να διατηρηθεί ή όχι κοινή θέση. Α επικεντρώσουμε την προσοχή μα στο, θέμα τη ε, ε διάσωση τη ζωή των υπολείπων και στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και α ξεκινήσουμε μια περίοδο νυφάλεια ε, συζήτηση και προβληματισμού ε, για το θέμα τα, τα ε, μελλοντική μα πολιτική απέναντι στην Κούβα. Όλα αυτά έχουν και προσθέμενη αξία. Το, το γεγονό ότι προέρχονται από έξι πολιτικέ ομάδε. Ξεκινάμε λοιπόν μια νέα περίοδο ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποτέ λοιπόν πια δεν θέλουμε ε, η ε, η δεξιά ε, στην Ευρώπη να υποκλίνεται στον ε, υπεριαλισμό των Γιάνκιδων, αν μου επιτρέπετε να πω την έκφραση. Ταυτόχρονα, οι σοσιαλδημοκράτε δεν θα πρέπει πλέον ε, να είναι συνένοχοι και να κλείνουν τα μάτια απέναντι στην κομμουνιστική δικτατορία. Ακριβώ διότι τα επιχειρήματα και από τι μεν και από του δε είναι ψευδή. Πρέπει όλοι να ενωθούμε απέναντι σε αυτού που σκοτώνουν του αγωνιστέ τη ελευθερία. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαφράγκα, ε, ο οποίο διαπραγματεύτηκε το κείμενο αυτό εξ ονόματο ε, του ΕΛΚ, επίση την εκπρόσωπο ε, του ΑΡΔΕ, τον κύριο Ρωμέβα εξ ονόματο τη ομάδα των Πρασίνων, τον κύριο Κασούσνικ, από του μεταρρυθμιστέ και συντηρητικού και όλου του συναδέλφου που συμμετείχαν σε, σε αυτέ τι δύσκολε περίπλοκε διαπραγματεύσει, αλλά που ελπίζω αύριο να στεφθούν από επιτυχία. Ε, με επιτυχία. Τέλος, ε, να ευχαριστήσουμε τον Προεδρεύοντα ε, του Συμβουλίου, τον κύριο Σαπατέρο, για την αμέριστη υποστήριξή του όσον αφορά την προώθηση αυτού του ψηφίσματος το οποίο συζητάμε σήμερα. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους. Κυρία Βέμπερ, εξ της ομάδας του Άλβε. Κύριοι συνάδελφοι, εκ μέρου τη πολιτική μου ομάδα, θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην ε, ε, οικογένεια του κυρίου Θαπάτο ε, Ταμάγιο, ο οποίο πλήρωσε ένα υψηλό τίμημα για τι πεπιτήσει του. Ο ακτιβισμό του για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτέλεσε πηγή έμπνευση για πολλού άλλου ακτιβιστέ και υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντό και εκτό τη Κούβα. Το ψήφισμα το οποίο προτάθηκε από, από αρκετέ πολιτικέ ομάδε εκφράζει τη βαθιά μα ανησυχία για τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Α είμαστε ειλικρινεί, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί και πολλοί ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, οι ειρηνικοί αντιφρονούντε και οι υπερασπιστέ της ειρήνης είναι φυλακισμένοι απλώ και μόνο επειδή θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα τη ελευθερία του λόγου και της, ε, του δικαιώματο του συναθρίζεστε. Ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει δεν μπορούν να εργαστούν γιατί η κυβέρνηση ασκεί έναν έλεγχο. Ε, την εποχή τη συζήτηση πολύ πολλοί πιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν απεργία πείνα. Και αυτό είναι λόγο ενσύστη ότι υπάρχουν ενδείξει γιατί υπάρχουν ενδείξεις για την επιδείνωση τη υγεία του κυρίου Γκυγέρμο Φαρίνια. Οι αρχέ τη ε, Κούβα ε, παραμελούν επαναλαμβάνουμε σε κλήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατούμενων και αυτό είναι ιδιαίτερο θλιβερό. Γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε ε, να, εγγυ... να εφαρμόσει όλου του μηχανισμού για να εγγυηθεί τι ζωέ εκείνων που προασπίζονται τα πλουραλιστικά δικαιώματα στην Κούβα εκ μέρους των Πρασίνων ο κύριος Ρεμέδα Ιρουέδα. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και μέσα της δικής πολιτικής ομάδας. Ε, ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας για την κατάσταση της Κούβα, το γεγονός αυτό είναι θλιβερό και χρειάζεται μια καταδίκη και κάτι παραπάνω, έναν προβληματισμό και μια υπενθύμηση. Θα πρέπει να ε, τονίσουμε την ανάγκη απελευθέρωσης όλων των ε, κρατούμενων για τις πολιτικές του παπαθήσεις στην Κούβα και σε, άλλες τις, και σε όλες τις άλλες περιοχές του πλανήτη. Νομίζω είναι αναγκαίο να το κάνουμε και είναι σημαντικό να το κάνουμε επίσης ανεξάρτητα επιμένω από τα κίνητρα, ε, από τα κίνητρα που μπορούν να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι αναγκαίο να ζητήσουμε την άμεση απελευθέρωση αυτών των κρατούμενων στην περίπτωση της Κούβας και να υπενθύσουμε την ευαίσθητη κατάσταση ορισμένων από αυτά τα πρόσωπα που συνεχίζουν, ε, συνεχίζουν την απεργία πείνας όπως είναι ο Γκυριέμο Φαρίνας. Επίσης, ε, βεβαίω υπάρχει ένας κίνδυνος να εκμεταλλευτεί κανείς πολιτικά την περίπτωση αυτή για άλλα θέματα για ζητήματα που μπορούν να είναι επικίνδυνα ή ολιστηρά. Και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι υπάρχουν πολλέ διαδικασίε εξέλιξη που είναι χρήσιμε, που λειτουργούν και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιπέσουμε στον πειρασμό να επιστρέψουμε σε παροχημένε ε, ε, περιόδους όπου χρησιμοποιούσαμε αυτή την ε, αξιοθρήνητη πολιτική του εμπάργου, και γνωρίζουμε τις επιπτώσεις της εάν δεν θέλουμε να επαναληφθούν καταστάσει όπως αυτή του Ολάντο Θαπάτα, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από κοινού, ούτε ώστε να αποφύγουμε ε, τέτοιου είδους ε, επαναλήψεις που ε, παραβιάζουν κατάφορα το κράτος δικαίου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κοσούσνικ για δύο λεπτά εξ ονόματος της ομάδας Ευχαριστώ πολύ είδηση για το θάνατο του Ορλάντα Ζαπάτα ε, μας ε, συγκίνησε πολύ και θα ήθελα να απευθύνω τα ε, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Γεννήθηκα το 1971, τότε που, που ήταν μια από τις σκληρές περιόδους της κομμουνιστικές στην χώρα μου, η πείρα της χώρας μου με την εγκληματική κομμουνιστική ιδεολογία ενέπνευνε στους ε, Τσέχους μεγάλη αλληλεγγύη απέναντι στον λαό της Κούβας. Λυπούμαθα πάρα πολύ για την είδηση αυτή που έφτασε από την Κίβα. Τόσα χρόνια μετά την επανάσταση της ε, Κούβας το σοσιαλιστικό ε, σλόγγαν εφαρμόζεται και δεν υπάρχει καμία ανοχή, καμία ανεκτικότητα. Ελπίζω ο θάνατος του Ορλάντο Ζαπάτα να μην ήταν μάταιος και να αφυπνήσει τον λαό της Κούβας. Στην χώρα μου το τελευταίο ε, θύμα της ε, κομμουνιστικού τρόμου πέθανε στην φυλακή Ελπίζω ότι ο Ζαπάτα θα είναι είτε το τελευταίο θύμα και θα ελευθερωθεί η Κούβα. Σας κάνω έκκληση διότι δεν θα υπάρξει πραγματική πρίοδο, πρόοδος απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουμένων και αρχή των μεταρρυθμίσεων για την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου ενώ δεν θα μπορούμε να αναθεωρήσουμε την κοινή θέση. Ο κύριος Μεγιάρ, δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ομάδα μου εκφράζει τη βαθιά τη λύπη για το θάνατο του κρατούμενου Ορλάντο Θαπάτα. Ε, ο κρατούμενο αυτό ε, ε, ε, ήταν ένα κρατούμενο και όπω σε κάθε περίπτωση ε, την ευθύνη για την υγεία του και τη ζωή του την έχει η κυβέρνηση. Και βεβαίω εκφράζουμε τη βαθιά μα λύπη. Εμεί όμω ε, δεν δεχόμαστε αυτή την εκμετάλλευση που γίνεται και τη σύνδεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα συζητάμε και αύριο θα ψηφίσουμε. Δεν το πράξαμε όμω με το πραξικόπημα στην Ονδούρα. Με, ε, ίσως είναι το μοναδικό κοινοβούλιο στον κόσμο που δεν συζητήσαμε και δεν καταψηφίσαμε ε, ε, το ε, πραξικόπημα στην Ονδούρα με τις δολοφονίες και, τις, ε, και τα βασανιστήρια που έγιναν. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με τη φιλοσοφία ότι δηλαδή ανάλογα με το πού γίνεται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τότε τοποθετείται το κοινοβούλιο. Πριν από, μία, πριν από εβδομάδες ανακαλύφθηκε στην Κολομβία ότι ο μεγαλύτερος ε, κοινό τάφο ε, στην Λατινική Αμερική. Από 2.500 έως 50.000 ε, υπολογίζονται τα, ε, τα θύματα. Το συζητήσαμε, το καταδικάσαμε. Τι γίνεται με τα θύματα των αμάχων στο Αφγανιστάν, τι γίνεται με τις διώξει στη Δυτική Ζαχάρα. Μα εκεί δεν, δεν είπαμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να είμαστε υποκριτέ. Είναι αλήθεια. Το βασικό είναι να υπάρξει μια ειλικρινή και άμεση σχέση και ένα διάλογο με την Κούβα για να, ε, ε, για να δούμε όλα τα ζητήματα και όλε τι πολιτικέ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κατάσταση στι φυλακέ. Αλλά ε, μια κατάσταση ισότιμη, σε, ισότιμη, σε ισότιμο διάλογο. Γιατί ε, ε, ε εμεί αυτή τη στιγμή έχουμε μια κοινή θέση προ την Κούβα ε, που δεν την έχουμε καμία άλλη χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. ούτε με τη λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα που αναφέρθηκε, ούτε με το Βιετνάμ. Γιατί, γιατί λοιπόν, γιατί με την Κούβα έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Και γιατί δεν έχουμε τη διαστάση απέναντι στη λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα. Ε, και απευθύνουμε και στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Πρέπει λοιπόν να απαντήσετε με, με ειλικρίνεια στην εξή ερώτηση. Θα ε, δοθεί τέλο στην κοινή θέση που για μένα αποτελεί ένα από τα πιο προφανή εμπόδια για να σημειωθεί πρόοδο σε ένα ειλικρινή διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία τη Κούβα με κοινά θέματα ε, που να αποτελούν ε, θέματα κοινού ενδιαφέροντο. Ευχαριστώ. Κύριος για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο θάνατος του κυρίου Σαπάτα και η σύλληψη του κυρίου Σάντσαθ ε, καθιστά σαφές ότι η σύνδεση της ε, ε, πολιτικής μας για την Κούβα θα πρέπει να συνδέεται ακόμα περαιτέρω όπως από το 1996 με τον εκδημοκρατισμό αυτής της χώρας. Οι εξαγγελίες του Κάστρο έχουν, περί εκδημοκρατισμού έχουν εξαλειφθεί. Οι πολίτες δεν απολάβουν εκείνων των ελευθεριών ε, που είχαν υποσχεθεί οι αδελφοί Κάστρο ε, και η κατάσταση είναι όπως ε, την εποχή του Πατίστα. Ε, οι πρωτοβουλίες αλλά και η ευημερία θεωρούνται ως κριτική του καθεστώτος. Η χαλάρωση του εμπάργου για κομπιούτερ και για software δεν ανταποκρίνεται στην αντίληψη που έχει η κοινή γνώμη, η ερμηνεία μάλλον των υποσχέσεων του Ομπάμα. Παρ' όλα αυτά θα συνεισφέρει στην καλύτερη οργάνωση της αντιπολίτευσης. Και ε, δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση της Κούβας γι' αυτό το λόγο να συνεχίσει την ε, απαγόρευση της ελευθερίας της έκφρασης. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πάψουμε να αγωνιζόμαστε για μια περαιτέρω χαλάρωση των απαγορεύσεων του κομμουνιστικού συστήματος. Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στον κύριο Βαλέσα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η τραγωδία του θανάτου του ε, φυλακισμένου στην Κούβα Ορλάντο Ζαπάτα είναι μια άλλη απόδειξη ότι το καθεστώς του Κάστρο αγνοεί ε, τελείως τις διεθνείς εκκλήσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και ε, να κλείσει την πολιτική αυτή της δίωξης αυτών που αγωνίζονται για τη δημοκρατική υπόθεση. Χρειάζεται πολιτική ε, διεθνής, αλλά πάρα πολλοί δεν θέλουν να μιλήσουν με τους αντιφρονούντες και δεν λαμβάνουν υπόψη την κοινή γνώμη στην Κούβα. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να καταβάλουμε μια κοινή προσπάθεια για να ασκήσουμε πίεση πάνω στο καθεστώς του Κάστρο και να ζητήσουμε την άμεση αποφυλάκηση αυτών που έχουν καταδικαστεί σε πολιετή φυλάκιση για τις απόψεις τους. Τα πρόσφατα χρόνια έχει μετριάσει τη θέση της Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει καταργήσει τις κυρώσεις κατά της Κούβας, νομίζοντας ότι έτσι η Κούβα θα ενθαρρυνθεί να ακολουθήσει πιο δημοκρατικά κριτήρια. Δυστυχώ, ο θάνατος του Ορλάντο Ζαπάτα δείχνει πόσο αφελής ήταν αυτή η πολιτική και αναποτελεσματική. Δεν πρέπει να την συνεχίσουμε. Αύριο θα ψηφίσουμε για το ψήφισμα μετά την σημερινή συζήτηση. Θα πρέπει να υπάρξει σαφής ε, προειδοποίηση ε, για την ε, καταδίκη αυτή από μέρους μας της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε αλληλεγγύη με τους Κουβανούς. Πρέπει να είμαστε η φωνή αυτών που δεν μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους. Ευχαριστώ κύριε Βαλέσα. Χέμιν Μπόσκοτ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η τραγική μοίρα του κυρίου Θαπάτο Ταμάγια οδήγησε παγκόσμια σε αγανάκτηση. Ε, ο κύριος Θαπάτα ήταν σε μια απελπιστική κατάσταση και μόνο με το θάνατό του έλπιζε ότι θα πετύχει κάτι. Ε, αγωνίστηκε κατά των συνθήκων κράτησής του και τελικά δεν μπόρεσε να εκφράσει την αναγανάκτησή του παρά μόνο με το θάνατο. Ποια ήταν τα εγκλήματα που είχε διαπράξει ο άνθρωπο αυτό για να καταλήξει στη φυλακή. Απλώ και μόνο ότι είχε μια εντελώ διαφορετική άποψη, αλλά αυτό δεν συνιστά έγκλημα. Ο θάνατο του Θαπάτα, ωστόσο, δεν συνιστά μεμονωμένη περίπτωση. Οι ψυχολόγοι και. Ο ψυχολόγος και δημοσιογράφος ε, Φαρίνια ξεκίνησε επίσης μια απεργία πείνας και θέλει να πετύχει την απελευθέρωση 26 άρρωστων κρατούμενων. Θα μπορέσει να το πετύχει ή θα πληρώσει και αυτός με το θάνατο του ένα υψηλό τίμημα τον φυλακίζονται άνθρωποι για τα ιδεώδη του αντιβαίνει ε, κατάφορα στη γενική διακήρυξη, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση για άμεση απελευθέρωση όλων των αντιφρονούντων. Μία κυβέρνηση δεν είναι το να κυριαρχεί το σκέπτεστε των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, έστω και αν είναι φυλακισμένοι, ε, μπορούν να σκέπτονται ελεύθερα. Δεν, είναι, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να προσπαθεί να καταργήσει κανείς κάτι τέτοιο. Η Κούβα έχει μια μακρά εμπειρία σε αυτό το επίπεδο. Μόνο μέσω του πολιτικού διαλόγου μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη. Γι' αυτό η κυβέρνηση της Κούβας είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο θάνατος του Θαπάτα ε, θα πρέπει να χρησιμεύσει σε κάτι. Ε, τουλάχιστον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα ελπίζουμε να προχωρήσει ούτε θα να υπάρξει μια βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται μόνο για ε, κρατούμενους συνείδησης ή αντιφρονούντες όπως είναι ο Θαπάτα, αλλά και για ακτιβιστές που παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κουβανική κυβέρνηση θα πρέπει να φροντίσει για τον πληθυσμό της. Δεν είναι δυνατόν επειδή φοβάται να συλλαμβάνει ανθρώπους και να τους μεταχειρίζεται ως εγκληματίες. Δεν μπορεί να αποστερήσει από τους πολίτες την ελευθερία της. Αυτό είναι ένα έγκλημα. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα σημαίνει ότι ε, καταδικάζουμε ε, τον, ε, τον, τον αδικαιολόγητο θάνατο του πολιτικού κρατούμενου Θαπάτα και την απελευθέρωση των υπόλοιπων κρατούμενων. Ελπίζω να ευαισθητοποιηθούν οι αρχέ τη Κούνα και τη Κούβα και να σημειώσουν πρόοδο προ μια πραγματική δημοκρατία. Στην Κούβα υπάρχει δικτατορία γιατί υπάρχουν κρατούμενοι συνείδηση, γιατί υπάρχει φόβο απέναντι στη συζήτηση, στην ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, υπάρχει ο φόβο προ την ελευθερία. και οι ιδέε δεν, είναι, δεν σκοτώνουν. Μπορεί να προκαλέσουν, να τρομάξουν, αλλά πάντα οδηγούν στη συζήτηση και ποτέ δεν πρέπει να οδηγούν στη φυλακή. Ε, κοιτάξτε, ε, δεν μπορούμε ε, να, ε, να απαγορεύσουμε το να σκέφτεται κανείς. Οι ιδέες λοιπόν και τα συναισθήματα τα οποία θέλουν ε, να καταπνίξουν η, η, η, η κυβέρνηση γίνονται νερό το οποίο πνίγει τελικά ε, τις κυβερνήσεις. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν. Όπως και στην περίπτωση του Μπατίστα που, και το, και το το οποίο έπεσε από την Επανάσταση. Τα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Και το Κοινοβούλιο μα αποκτά αξιοπιστία όταν αντιδρά το ίδιο έντονα απέναντι σε όλε τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού. Στο Αφγανιστάν, στην Παλαιστίνη, ε, στην ε, χώρα των Βάσκων, ε, στην Κολομβία, παντού. Αυτή πρέπει να είναι η δέσμευσή μα. Τουλάχιστον είναι η δική μου. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάο. Το λόγο έχει ο κύριο Πορέμπα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όλοι εδώ συμφωνούμε νομίζω ότι ε, οι διεφθαρμένοι ε, δικτάτορες δεν επιτρέπουν καμία αλλαγή στην Κούβα. Ε, τουλάχιστον οι αδελφοί Κάστρο έχουν καταστρέψει την ελευθερία των πολιτών και τους έχουν στερήσει κάθε ευπρεπή ζωή, κάθε ευπρέπεια στη ζωή τους πρέπει να έχουμε ένα ρόλο εδώ, θα πρέπει να δράσουμε για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη προϋπόθεση για ένα διάλογο με την Κούβα. Πρέπει να υποστηρίξουμε την δραστηριότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων την πρόσβαση στο ε, διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης οι διατλαντικοί δεσμοί μπορεί να είναι σημαντικοί εδώ, γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τη Ουάσιγκτον. Μαζί μπορούμε να ετοιμάσουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ε, Κούβα. Δεν πρέπει να δεχθούμε το status quo, αλλά να επιβάλλουμε μια, ε, ένα όραμα δημοκρατίας. Hilda Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση για άλλη μια φορά δείχνει ότι ε, χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και σταθμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, από τη μια ε, υπάρχουν ορισμένοι που δεν θέλουν να ε, κατα, καταδικάσουν την κατάσταση στην Ονδούρα, ε, όπου και εκεί ε, υπήρξαν πολλά θύματα και τώρα ξεκινούν διαπραγματεύσεις σύνδεσης με μια κυβέρνηση που προήλθε όπως όλοι ξέρουμε πώς προήλθε. Βεβαίω όλοι εκφράζουμε τη λύπη μα για το θάνατο ε, του ε, Θαπάτα από απεργία πείνα. Αλλά δεν μπορούμε να, ε, να ξεχνάμε ε, ότι εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη στάση απέναντι στην Κούβα με τρομερέ συνέπειε από όλε τι απόψει. Μην ξεχνάμε ταυτόχρονα τους πέντε κουβανούς που είναι φυλακισμένοι σε φυλακές των Ηνωμένων δεν μπορούμε λοιπόν ε, να, παρά να ζητήσουμε ε, την σύναψη ανοιχτών σχέσεων με την ε, Κούβα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε, προλαβαίνουμε να αποσύρουμε την κοινή στάση για να βελτιωθούν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κούβα. Αυτό περιμένουμε από την Ισπανική Προεδρία. Ευχαριστούμε και το λόγο του κύριο Σόνι και δύο λεπτά. Ναι. Θυμόμαστε ακόμα τι είπε ο Φίδελ Κάστρο, σοσιαλισμός ή θάνατος. Αλλά τώρα έχουμε μόνο θάνατο και καθόλου σοσιαλισμό. Έχουμε το θάνατο του Ορλάντο Ζαπάτα, ε, του πατριώτη Ορλάντο Ζαπάτα Ντεμάγιο και όλα αυτά έθεσε σε κίνδυνο την ιδέα του σοσιαλισμού. Πηγαίνοντα η Κούβα νομίζω ντροπιάζει όσους βρίσκονται στην αριστερά. και εγώ επίσης αισθάνθηκα ντροπή όταν έγινε μια επίσκεψη στην Κούβα, όταν προσφέρθηκε συνεργασία, αλλά δεν οργανώθηκαν συναντήσεις με αντιφρονούντες. Πρέπει να το ξεχάσουμε, διότι δεν υπήρξαν ποτέ δημοκρατικές εκλογές στην Κούβα και υπάρχουν οι αντιρρησίες συνείδησης είναι ακόμα στην φυλακή. Ποια πολιτική απέναντι στην Κούβα. Η προϋπόθεση είναι βεβαίως η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, η εξάλληψη της λογοκρισίας, η αποκατάσταση των ε, πολιτικών και δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των πολιτών. Πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό το θέμα. Υπάρχουν ε, διαφορετικοί τρόποι να ελευθερωθεί από το δικτατορικό καθεστώς. Υπάρχει ο τρόπος του διαλόγου και υπάρχει και ο τρόπος που ακολούθησε η Ρουμανία όπου το σενάριο ήταν τελείως ε, διαφορετικό και δραματικό. Θέλουμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο σενάριο. Τι δρόμο θα ακολουθήσει η Κούβα. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει ενεργά να συμβάλλει στο να γίνει η Κούβα χώρος ελευθερίας και δημοκρατίας και αυτή πρέπει να είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, ευχαριστώ Σονίκ, τώρα Χόιτ, ευχαριστώ, εκφράζω τα συλληπιτήρια για το θάνατο του Ορλάντο Ζαπάτα Ντεμάγιο ε, και την συμπάθειά μου για τους αντιφρονούντες που άρχισαν ε, απεργία πείνας για αλληλεγγύη. Θα πρέπει να ζητήσουμε ανεφόρον την απελευθέρωση των, ε, των κρατουμένων συνείδησης. Υπάρχουν πάρα πολλοί κρατούμενοι και οι οποίοι μας ανησυχούν για τον, την κράτηση και τον ξυλοδαρμό του Ντάσο Φερέρ στην Αβάνα. Για 19 χρόνια δεν υπήρξε πρόσκληση ε, στην Κούβα. Πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση της Κούβας να ε, θέσει ε, για ημερομηνία για την επίσκεψη του Νόβακ, του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τους βασανισμού. Πάντοτε έχουμε αντιτεθεί στο εμπάργο των Ηνωμένων Πολιτειών, το εμπορικό αποκλεισμό και νομίζω μέτρα εγκρίθηκαν από τον πρόεδρο Ομπάμα ούτω ώστε οι κουβανοί Αμερικανοί ε, να ταξιδεύουν πιο ελεύθερα και να στέλνουν περισσότερα εμβάσματα στην πατρίδα τους. Έχουμε την κοινή θέση για πολιτικό διάλογο μεταξύ Κούβας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποκατάσταση ε, μιας αναπτυξιακής συνεργασίας. Ε, χαιρετίζω το γεγονός ότι η BBC έχει τώρα ελεύθερη πρόσβαση στην Κούβα, αλλά εκφράζω την απογοήτευση διότι στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Εθνών η Κούβα δεν δέχθηκε τις συστάσεις να επικαιρώσει τις δύο συνθήκες δηλαδή που θα επιτρέψουν την ελεύθερη επίσκεψη των φυλακών. Εσείς και όλοι μας που έχουμε επισκεφθεί την Κούβα θα πρέπει να επιμείνουμε ότι ε, χρειαζόμαστε αυτές τις προόδους στην Κούβα. Ε, πέρσι υπήρξε μια επίσκεψη υφυπουργού στην Κούβα και θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε το ίδιο, χωρίς όρους. Τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Λουί Μισελ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, κύριε ε, Υπουργέ, ο θάνατος του Ορλάντο Ζαπατάη είναι απόδειξη της απόγνωσης την οποία μπορεί να οδηγήσει η έλλειψη ελευθεριών πρέπει να καταγγείλουμε την φυλάκιση τόσων ατόμων ε, στις φυλακές. Ε, δεν μπορούμε ε, να δεχθούμε την αυθαιρεσία ενός καθεστώτος που στερεί τις βασικότερες ελευθερίες από τους πολίτες. Αλλά πρέπει να έχουμε έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος είναι η έκφραση πιο απτή των ευρωπαϊκών μας αρχών. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας είναι περίπλοκες και συχνά βασίζονται σε έλλειψη κατανόησης που οδήγησε σε ακαμψίες σοβαρές που υπονομεύουν τις προοπτικές ενός πολιτικού διαλόγου και τις προόδους ενός τέτοιου διαλόγου. Βρίσκεται σε καμπή της ιστορίας της η Κούβα και είμαι πεπισμένος ότι θα ήταν σφάλμα να μην υποστηρίξουμε ακόμα και τις προόδους τις περιορισμένες που τρέφονται από ιδιαίτερη ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίσως η μοναδική πολιτική εξουσία που είναι ικανή να πείσει τους κουβανούς ότι η απομόνωσή τους είναι αυτοκτονησιακή και θα τους οδηγήσει σε μοίρα δραματική. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την ευθύνη που έχουμε να συνεχίσουμε το διάλογο χωρίς να ε, αποκλείσουμε κανέναν αλλά ε, καμιά φορά υπάρχουν διπλοί κανόνες, διπλά μέτρα και σταθμά. Τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Μιγκάλσκι για ένα λεπτό. Ε, κύριε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ελευθερία στην ε, Κούβα θα κατησχίσει, θα υπάρξει δημοκρατία και ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει την ουσία να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση, αλλά θέλει να βοηθήσει το κουβανικό πληθυσμό αυτή τη στιγμή γίνει μια πολιτική αλλαγή. Και οι εμπειρίε από άλλε χώρε μα έδειξαν ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της μελλοντικά να μην ε, υπάρξει η κατάσταση την οποία περιγράφει ο Πολωνό συγγραφέας Μαγιαρόφσκι. Δηλαδή, οι αντιφρονούντες να μην γίνονται μελλοντικά αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ο κύριος Μιστάλκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να δισταθεί μια ανθρώπινη ζωή ε, λυπούμε για κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται και πραγματικά συμμερίζουμε τη θλίψη σας για το θάνατο του αντιφρονούντος. Ε, δυστυχώς θα πρέπει να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα πρόσφατα κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντρική Ασία. Είπα τότε ότι, αυτό, ότι, υπήρξε, ότι ήταν ένα σφάλμα να μην ε, σέβεται κανείς τις ιστορικές και πολιτιστικές παραδόσεις συγκεκριμένων χωρών και να μην ε, σέβεται κανείς τα θετικά αποτελέσματα που έχουν πετύχει οι χώρες αυτές. Και αυτό ισχύει και για την Κούβα. Για να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Κούβα θα πρέπει να έχουμε έναν ισότιμο διάλογο στον οποίο ε, συνενούν οι κουβανικές αρχές. Ε, θα πρέπει επίσης να βοηθήσουμε στη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης στην Κούβα. Παρά τις οικονομικές ε, δυσχέρειες, η Κούβα είναι πάντοτε πρόθυμη να βοηθήσει τις άλλες χώρες, για παράδειγμα στην περίπτωση της ε, καταστροφής στην ΑΙΤ. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε καταδίκες. λεπτά. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το γεγονός ότι σήμερα και κυρίως αύριο όταν θα ψηφίσουμε θα ε, γράψουμε μια νέα σελίδα ε, γεμάτη αξιοπρέπεια ε, στην ιστορία του Κοινοβουλίου. Γιατί για μία φορά, αφήνοντα στην άκρη τι αμοιβέ προκαταλήψει και το γεγονό ότι ανήκουμε σε διαφορετική διαφορετικούς πολιτικού σχηματισμούς ναι, ερχόμαστε ε, να ενωθούμε όλοι απέναντι στο ύψιστο μυστήριο του θανάτου ενός ανθρώπου και να ε, προσυπογράψουμε την αλήθεια. Γιατί τι λέμε τελικά σε αυτό το ψήφισμα. Αναφέρουμε πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται στοιχειώδη, μπορεί να φαίνονται προφανή, αλλά στην ουσία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γράφουμε ότι στην Κούβα δεν υπάρχει ελευθερία. Γράφουμε ότι στην Κούβα δεν υπάρχει δημοκρατία. Γράφουμε ότι, ε, ε ότι η ζωή είναι αγαθό και δεν θα πρέπει κανείς να την αφαιρεί Όλα αυτά που μπορεί να φαίνονται προφανή. Αλλά έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να ξεπεράσουμε ε, και οι μεν και οι δε τι προκαταλήψει μα και να αναγνωρίσουμε ένα γεγονό το οποίο δεν προσβάλλει ε, καμία πολιτική πεποίθηση. Απλά και μόνο μα οδηγεί στο να αναγνωρίσουμε αυτό το στοιχειώδε στοιχείο αλήθεια πάνω στο οποίο και μόνο στηρίζει το διάλογο. Εμεί λοιπόν δεν πρέπει ε, ε, ε, να, να, μην, να, μην προωθούμε το διάλογο με την Κούβα. Αλλά αυτός ο διάλογο πρέπει να είναι αληθινό. Άρα πρέπει να ξεκινά από την αλήθεια. Και ε, άρα από το γεγονό ότι, ο, άνθρωπος πρέπει να γνωρίζεται ω κεντρικό στοιχείο τη ελευθερία. Και ότι μαζί με τι εκδηλώσει συμπάθεια απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε η κυβέρνηση Κάστρο να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παραμικρή υποχώρηση. και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αποτελούν ένα, ε, ένα σημαντικό στοιχείο και όχι δευτερεύον. Λοιπόν, ε, ε, αξιοποιήσαμε την ευκαιρία, αλλά δεν το έπραξε η ύπατο εκπρόσωπο. Και σήμερα το πρωί υπενθυμίσαμε ότι το Κούμπα Λίμπρε δεν είναι ένα κοκτέιλ. Είναι η κραυγή που βγαίνει από τα βάφη τη καρδιά μα. Γιατί θέλουμε τη δημοκρατία και θέλουμε την ελευθερία στην Κούβα. Merci, Ευχαριστούμε κύριε Μάουρο. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μούνη Ντεουρκίσα. Σα ευχαριστώ, ε, κυρία Πρόεδρε. Οι σοσιαλιστέ στην Ισπανία εκφράζουμε τη βαθιά μα λύπη για το θάνατο του Ορλάντο Θαπάτα και για την κατάσταση ε, των ε, κρατούμενων συνείδηση στην Κούβα και ζητούμε αποφασιστικά την απελευθέρωσή του. Ο θάνατο του Θαπάτα είναι ένα πολύ λυπηρό γεγονό, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να αποτελέσει αφορμή έτσι ώστε για να, να αφήσουμε ε, ε, ε, τις συζητήσεις τις γενικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μιλήσουμε με τις αρχές της Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την αλλαγή της κοινή θέση που μας εμποδίζει να έχουμε οποιοδήποτε διάλογο με τις αρχές της Κούβας. Γιατί τελικά οι αρχές της Κούβας είναι αυτές που έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις συνθήκες στο νησί. Η κοινή θέση βεβαίως δεν είναι πλέον κοινή γιατί μεγάλο μέρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί διμερείς σχέσεις, ενεργές διμερείς σχέσεις με την Κούβα και ε, ε, η κοινή θέση αποτελεί εμπόδιο απέναντι σε οποιαδήποτε δυνατότητα θέσπιση ε, πολιτικού διαλόγου. Και γι' αυτό δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει το διάλογο αυτό με βάση τι αρχέ που διαπνέουν την κοινή εξωτερική πολιτική και τι αρχέ τη πρόθεση τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κοινή θέση είναι ένα παροχημένο μέσο που ενεκρίθη από 15 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση τον περασμένο αιώνα. Τώρα όμω είμαστε 27 κράτη-μέλη. Η κατάσταση στον κόσμο άλλαξε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν διάλογο με την Κούβα για λεπτά και ευαίσθητα ζητήματα όπω η μετανάστευση. Ε, Επίση, ε, ε, ε, έγινε δεκτή σε διάφορου διεθνεί οργανισμού η Κούβα με βάση τι αρχέ διαλόγου και δημοκρατία και τώρα εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε ένα μέσο το οποίο θα μα επιτρέψει να προωθήσουμε αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε, αυτό που αποτελεί την ουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τι αρχέ δημοκρατία. Ο διάλογο με την Κούβα δεν είναι πολυτέλεια. Ε, ε, ε, ε, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε αναπτύξει σχέσεις με χώρες που δεν πληρούν ούτε κατελάχιστον τις αρχές του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Μόνο ο διάλογος και μηχανισμό μηχανισμός συνεργασίας και δέσμευσης μέσω των διεθνών φόρων θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει κάτι από την Κούβα. Και αυτοί που αρνούνται το διάλογο δεν θέλουν τελικά να υπάρξει δίκαιη λύση απέναντι σε αυτούς που θέλουμε να υπερασπιστούμε, στου αγωνιστές της δημοκρατίας. Όμως η κυβέρνηση της Ισπανία μέσω του δημοκρατικού διαλόγου ε, έδειξε ότι είναι αποτελεσματική η εξωτερική τη πολιτική και πέτυχε την απελευθέρωση σημαντικού αριθμού ε, πολιτικών κρατούμενων. Τελειώνω. Ε, ο Δον, ο Κιχώτης είπε ότι αυτοί που τιμωρούνται με τα γεγονότα δεν χρειάζεται να τιμωρούνται και με τα λόγια. Α αφήσουμε λοιπόν τα λόγια και α αρχίσουμε να εργαζόμαστε συγκεκριμένα σε συνεργασία με τι αρχέ τη Κούβα. Γιατί αυτό χρειάζονται και οι ίδιοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και όχι οι ρητορικέ καταγγελίε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ραμόν Τρεμόσε, η Μπαλτσέλς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στη, στη μαύρη άνοιξη της ε, Κούβας το 2003, 75 αντιφρονούντες ε, φυλακίστηκαν ως ε, κατάσκοποι των ΉΠΑ. Τότε είχε φυλακιστεί και ο Ολάντο Θαπάτο. Οι γυναίκε ε, των ε, κρατουμένων δημιούργησαν τις Ντάμα Δεμπλάνκο, τις κυρίες με τα λεφτά που έλαβαν το βραβείο Ζαχάροφ. Σα υπενθυμίζω ότι το καθεστώ του Κάστρο δεν έδωσε το 2005 στι γυναίκε στις κυρίες με τα λευκά για να έρθουν εδώ να λάβουν το βραβείο του. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Κούβας αναγνωρίζει ότι στη χώρα αυτή υπάρχουν περί τους 200 πολιτικούς κρατούμενους. 22 από αυτούς είναι δημοσιογράφοι. Κούβα είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο στον αριθμό των φυλακισμένων ε, δημοσιογράφων. Μετά ε, το Ιράν με 52 και ε, τις Κίνες με 44 άτομα. Ο κύριος Σταπάτα δημιουργήθηκε, χαρακτηρίστηκε ως κρατούμενος συνείδησης, ξεκίνησε απεργία πείνας 85 ημερών πέθανε στι 23 Φεβρουαρίου, 85 μέρε μετά το ξεκίνημα τη απεργία πείνα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη με την οικογένεια του Θαπάτα και να εκφράσει την μεγάλη ανησυχία του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα. Το σώμα μα πρέπει να δώσει ένα σαφέ μήνυμα στο καθεστώ του Κάστρο, ιδιαίτερα στα πλαίσια τη Ισπανική Προεδρία μια προεδρία που σίγουρα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο δραστήρια στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Κούβα. Αγαπητοί συνάδελφοι, εν τέλει, με την ευκαιρία αυτή θέλω να ζητήσω την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στην Κούβα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Τρομόζα. Ο κύριος Μιλάν Μον είναι ο επόμενος ομιλητής για δύο λεπτά. Μεταξύ των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, βασική θέση έχουν η δημοκρατία και η πρόσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το άρθρο 21 της Ένωσης εφαρμόζεται και στις σχέσεις της με την Κούβα. Δυστυχώς, τα τελευταία πέντε χρόνια η δράση του Συμβουλίου φαίνεται ότι περιορίστηκε κατά βάση στην επιθυμία διόρθωσης της θέσης που είχε δηθεί τα προηγούμενα έτη, ιδιαίτερα το 2003, μετά από μια σκληρή καταπίεση στην Κούβα. Έκτοτε ε, το Συμβούλιο Κτάργησε τα μέτρα του 2003. Υπήρξαν επισκέψεις υπουργών επιτρόπων στην Κούβα. Ξεκίνησε ένα πολιτικός διάλογος ε, σφαιρικός, όπου θύμισε ο κ. Λόπεθ Γκαρίγκα σε υψηλό επίπεδο. Ο αρχηγό κράτου ενό κράτου μέλου πήγε πρόσφατα, επισκέφθηκε πρόσφατα την Κούβα. Δυστυχώ οι Ευρωπαίοι πολιτικοί που πήγαν στο νησί δεν είχαν ούτε μία στιγμή να συναντηθούν με του εκπροσώπου των αντιφρονών του που αισθάνονται ότι είναι στο περιθώριο. Όλο αυτό το χρόνο, το, την περίοδο η καταστολή στην Κούβα συνεχίστηκε. Δεν υπήρχαν μεταρρυθμίσει, δεν υπήρξαν αλλαγέ. Συνεχίστηκε ωστόσο ο διάλογο μαζί του. Τώρα όλοι έχουμε να τριχιάσει από τον φρικτό ομό του Ορλάντο Θαπάτο. Όπως γνωρίζετε, κάποια, μια κυβέρνηση όπως και η Ισπανική επανέλαβαν ότι θέλουν να καταργήσουν την κοινή θέση που λέει κάτι πολύ λογικό. Η υποστήριξη στην μεταβατική ε, στη δημοκρατική μετάβαση. Η υποστήριξη των βασικών αρχών, δηλαδή το άρθρο 21 της συνθήκης. Τελειώνω με δύο παρατηρήσεις. Η κοινή θέση ε, περιλαμβάνει διάλογο, είναι προφανές. Επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και από τους υπουργού τον 27 τον Ιούνιο του 9. Δεύτερον, δεν μπορεί η προτεραιότητα να είναι αλλαγή της κοινή θέση, αλίμονο, αλλά να ζητήσουμε την άμεση και πλήρη, χωρίς όρους, απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Η Κούβα, στην Κου, η Κούβα και η Λατινική Αμερική είναι για μένα δύση. Τα χαρακτηριστικά της δύσης είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Μια τελευταία παρατηρήση. Να υπενθυμίσει το Συμβούλιο ότι στα συμπεράσματά του τον Ιούνιο του 9 περιλάμβανε ε, φράση ότι ο διάλογος με τις αρχές της Κούβας ήταν υπό την αίρεση των εξελίξεων και της προόδου στην ε, προάσπιση των ε, πολιτικών ελευθεριών. Μπορείτε να βεβαιώσετε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Μιλάν. Ο κύριο Μάση Πιντάλγο για λεπτά. Η ιστορία θα με αθώσει. Αυτά τα είπε ένας νέος δικηγόρος ο οποίος έγινε εξεργέθηκε προσπατεύοντας τον λαό του κατά της τυραννίας και κατά του ε, αμερικανικού εμπάργου. Με, την ίδια δήλωση ωστόσο και το κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο χώρο ελευθερίας και δημοκρατίας στον κόσμο καταδικάζει την δικτατορία που πλήττει τον λαό της Κούβας. Η καταπίεση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο νησί η αονελέητος τρόπος αντιμετώπισης των πολιτικών κρατουμένων, η περιφρόνηση των εξορίστων, η κρίση της ιστορίας είναι σαφής με αυτό το ψήφισμα βουλευτές όλων των ιδεολογικών θέσεων στεκόμαστε δίπλα στους κουβανέζους που αγωνίζονται. Πρέπει να αποφύγουμε πάση φυσία την ομή καταπίεση που υφίστανται από την, και από την λεγόμενη κοινή θέση. Στον τελευταίο στίχο του Ριβέρο έλεγε ο ποιητής αυτός ε, η περιφρόνηση αυτή δεν δεν περιβάλλεται, δεν ε, στηρίζεται στην, ε, ε από, στην βεβαιότητα. Η, βεβαιότητα οδηγεί στην καταστροφή της πατρίδας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο θα δώσω τώρα στον κύριο Προβέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μια ακόμα φορά, η συμπεριφορά και οι επιλογέ του κομμουνιστικού καθεστώτο τη Κούβα θέτουν το Κοινοβούλιο ενώπιον ενό διλήμματο. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί ο διάλογο με το καθεστώ αυτό. Εδώ και έτη το Κοινοβούλιο ζητά από τις κουβανικές αρχές να υπάρξουν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το πέρασμα της εξουσίας ωστόσο από τον Φιντέλ Κάστρο, τον αδελφό του Ραούλ, δεν έφερε ούτε μεταρρυθμίσεις ούτε απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Ο θάνατος στη φυλακή του Ορλάντο Σαπάτα μετά από 85 μέρες απεργίας πίνες δείχνουν την ιδεολογική και κατασταλτική φύση του καθεστώτος. Σε 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε 145 εκατομμύρια ευρώ ε, την ε, ανοικοδόμηση και τις μεταρρυθμίσεις στην Κούβα. Δεν είναι νομίζω εξαιρετικά τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης αυτής. Αντίθετα, η χρηματοδότηση αυτή βοήθησε στην διαιώνιση της τυραννίας. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει να διακδικήσουμε οι σχέσεις με την Αβάνα και η αναπτυξιακή βοήθεια να συνδέονται με συγκεκριμένα επαληθεύσιμα μέτρα βελτίωσης και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου για όλους τους πολίτες της Κούβας και την άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Δεν θέτουμε ζητούμε και απαιτούμε αλλαγέ από ένα από τα πιο καταπιεστικά καθεστώτα του πλανήτη που είναι ο επίγονό μια ιτημένη τη ε, ιδεολογία τη ιστορία και που έχει το μέλλον τη είναι εξαφάνιση. Ευχαριστώ κύριε Προβέρα. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Γκάλερ θα είναι ο πρώτος ομιλητής. Wir sollten den Menschen in Kuba, aber auch dem Regime ein konkretes Angebot machen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 Πριν από τον Κάστρο. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Ο κύριος Φερέρα έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, θρυνούμε για το θάνατο του Ορλάντο Ζαπάτα. Λυπούμαστε που χρειάστηκε να φτάσει μέχρι το τέλος για τους λόγους που τον υποκινούσαν. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ο λόγος αυτού του θλιβερού γεγονότος να επιτρέπει ε, διαμαρτυρίες κατά της Κούβας όπως και αν κρίνουμε την επιλογή του κουβανικού λαού πρέπει να δεχθούμε τη δυνατότητα για αυτό το λαό να αποφασίζει για την τύχη του. Καταδικάζουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια παρεμβολής όπως τον αποκλεισμό στον οποίο υπόκειται εδώ και 1,5 αιώνα περίπου η Κούβα πιστεύουμε ότι η λογική αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι η εξομάλυση των σχέσεών της με την Κούβα, να, πάψει να εφαρμόζει διακρίσεις κατά της Κούβας και του λαού της. Και δεν μπορούμε να δεχθούμε επίσης την υποκρισία που διαπιστώνουμε ε, στα λόγια πολλών βουλευτών. Καταδικάζουμε επίσης την πολιτική των δύο μέτρων και σταθμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Λόπετ Τόριτς, ο επόμενος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απευθύνομαι προς την μητέρα του Ελλάδος Απάντα και τους συντρόφους του στην ε, μάχη για την ελευθερία στην Κούβα. Να τους πω ότι δεν είναι μόνοι. Το Κοινοβούλιο σήμερα με το ψήφισμα αυτό, ως Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, για την οποία ευχαριστώ τους συντάκτες, ιδιαίτερα δε τα κόμματα που υπέγραψαν το ψήφισμα αυτή, το Κοινοβούλιο έλεγα υψώνει τη φωνή ενωμένο κατά της απομονωμένης και σε αυτή τη δημοκρατία. Σήμερα έχουμε, βρισκόμαστε μπροστά στην ε, πρώτη μέρα της ε, θανατικής καταδίκη του καθεστώτο αυτού. Καταδικάζουμε τον θάμαντο, ξεκάθαρα τον θάνατο του Ορλάντο Ζαπάτα, θέλω να το πω στη μητέρα του. Πέραν αυτού, ωστόσο, ζητούμε την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων στο νησί χωρί όρου. Θα επαγρυπνούμε για την εξέλιξη τη κατάσταση, για την συνεχή παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο νησί. Ω Ευρωπαϊκό Λογικό Κόμμα, αλλά και άλλε πλευρέ, όπω άκουσα, θα αγωνιστούμε για να διατηρηθεί η κοινή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα δώσουμε μηνύματα σύγχυση, αλλά έναν σαφή δρόμο για να επιτύχουμε το όνειρό μα να δούμε μια δημοκρατική Κούβα η ύψιστη θυσία του Ορλάντο ταράσει τη συνείδηση του καθενός. Θέλουμε σε μια ελεύθερη Κούβα σύντομα να γιοτάσουμε, να, να, να, να θυμηθούμε τον θάνατό του. Ε, Κυρίες και κύριοι, για μας ε, νομίζω ότι είναι αρκετά απλό το να μιλάμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλα μέρη του κόσμου και για το ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν για τις πεπιθήσεις τους. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Ο κύριος ε, Θαπάτα με την απεργία πείνας έχασε τη ζωή του και υπάρχουν και άλλοι κρατούμενοι οι οποίοι και αυτοί ε, κάνουν απεργία πείνας. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Αναφέρθηκε αφενός ότι δεν πρέπει να μιλάμε με την Κούβα γιατί δεν δεχόμεθα το καθεστώς της. Από την άλλη ο κύριος Φερέρα Σήμερα είπε και κακός ότι εδώ ε, επικρατεί φαρισαϊσμός και ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους Κουβανούς να αποφασίσουν μόνοι τους. Η ελευθερία να αποφασίσουν ε, οι άνθρωποι μόνοι τους ε, δεν ισχύει όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι λοιπόν απόλυτα σωστό ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν κατατεθεί και από τον κύριο Γκάλα να συζητηθούν σε βάθος για να δούμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε έτσι ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονται σε όλα τα μέρη του κόσμου να τα προφυλάσσουμε για να βοηθούμε και τους ανθρώπους στα διάφορα σημεία του κόσμου. Ευχαριστώ κυρία Μέσνερ. Λυπούμαστε για το γεγονός ότι στον πίνακα αναφέρθηκε άλλο όνομα και όχι το δικό σας. Ο κύριος Όμπεν Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα βρισκόμαστε υπό την τραγική ε, εντύπωση και απήχηση του θανάτου του κ. Σαπάτα και μιλάμε για την Κούβα. Πρέπει να ξέρουμε ότι η εικόνα ε, που ισχύει σήμερα προέρχεται από τις εποχές όπου υπήρχε το πρότυπο του εχθρού. Ο κακός ο Κουβανός, ε, ο οποίος συνεργάζεται με την Σοβιετική Ένωση και από την άλλη ο καλός ο Κουβανός, ο οποίος διώχνει τη CIA και τον υπεριαλισμό. Φαίνεται όμως ότι ο κακός ε, καταπιάζει τους ανθρώπους και ο άλλος ο καλός είναι εκείνος ο οποίος έφερε τη χώρα ε, στο χείλος του λοιμού. Σήμερα λοιπόν, αν θέλουμε να έχει νόημα ο θάνατος του Θαπάτα, γενικά αν θέλουμε ο θάνατος να έχει νόημα, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε το τι ακριβώς συνέβη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να, καθαρίσει, να καθορίσει ένα σαφή δρόμο και να απελευθερωθεί από τις υποθήκες παρελθόντος. Να μην εφαρμόζουμε προθύστερα σχήματα, να ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύντομα να μπορούμε να μιλάμε για μια ελεύθερη Κούβα και να μπορεί ο, ο κόσμος και ο λαός να ζει σε ελεύθερη δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Ομπερμάγερ. Ο κύριος Βάτσερ έχει το λόγο τώρα. varit gällande οι Ηνωμένε Πολιτείε κρύβονται πίσω από όλα αυτά και αυτό επηρέασε το λαό της Κούβας επιβάλλοντας φτώχεια και δυστυχία. Νομίζω ότι πολλοί γνωρίζουν ότι η Human Rights Watch παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Κούβα. Στην έκθεσή της ανέφερε ότι πρέπει να σταματήσει το εμβάργο και να δοθούν έξι μήνες στους δικτάτορες στην Κούβα να ελευθερώσουν όλους τους κρατούμενους και να το πράξουν θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα πιο έξυπνο εμπάργο. Ένα εμπάργο που έχει εφαρμοστεί πολλές φορές πάγωμα των ε, περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύσεις στις μετακινήσεις και στα ταξίδια τα μεγαλύτερα δημοκρατικά κράτη και οι Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να υποστηρίξουν μια τέτοια πολιτική. Και θα θέλαμε να μας πει ο Υπουργό τι πιστεύει για αυτή την πρόταση της Human Rights Watch. κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς ε, λοιπόν ε, τον αγώνα ε, κατά τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, τον αγώνα αυτό πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε ω προτεραιότητα. Ο Ορλάντο Θαπάτα πέθανε γιατί διαμαρτυρήθηκε και άλλοι επίσης ε, διαμαρτύρονται. Υπάρχουν και άλλοι 25 άνθρωποι που βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση υγείας. Δεν αρκεί λοιπόν τους, ε, στους κρατόμενους ε, να προσφέρει κανείς άσυλο όπως το πράττει η Ισπανική κυβέρνηση. Η απελευθέρωση των κρατουμένων είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και κατά τα άλλα θα ήθελα να παρακαλέσω τον αρμόδιο επίτροπο η Επιτροπή να έρθει σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Κούβας και ο Ερυθρός Σταυρός να αποκτήσει την ευκαιρία να επισκεφθεί τους ε, κρατουμένους. Ε, κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τους κρατουμένους και θα συνέβαλε και στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ κύριο Ζαμπόρσκα. Τελευταία ομιλήτρια η κυρία Ούχτμαν. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ είμαι υπέρ τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου και στην Κούβα. Ο θάνατο του κυρίου Θαπάτα είναι η κραυγή αγωνία ενό ανθρώπου που βρέθηκε σε απαράδεκτη κατάσταση. Εγώ λοιπόν εύχομαι εμεί οι Ευρωπαίοι να ε, παρουσιάσουμε μία καθαρή γραμμή για την διαφύλαξη του χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ ανεξάρτητα από το καθεστώ στο οποίο ζούμε. Πολύ ωραία. Εξ του Συμβουλίου θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λόπες Γκαρίντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση που έγινε για το θέμα της κατάστασης των κρατούμενων, των πολιτικών κρατούμενων στην Κούβα λόγω του θανάτου ενός από αυτού του θα Θαπάτα επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένας εξαιρετικά υψηλός βαθμός σύμπτωσης των θέσεων μεταξύ βουλευτών από όλες τις πολιτικές ομάδες, όπως θα αποδειχθεί, είμαι πεπισμένος, αύριο στην ψηφοφορία για τα ψηφίσματα που θα προκύψουν από τη ζήτηση αυτή και που θα ακολουθούν κατά βάση μια γραμμή που συμπίπτει με αυτή που έχει το Συμβούλιο και η Επιτροπή και όλα τα όργανα της Ένωσης. Κάτι που σίγουρα ενισχύει την Ευρωπαϊκή Ένωση στον αναγκαίο διάλογο με την Κούβα και με στόχο να προχωρήσει και να βελτιωθεί η κατάσταση για τον κουβανικό λαό. Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πως είναι αναγκαίο να βγούμε υψώνοντας τη φωνή μας οπουδήποτε υπάρξει παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό είναι μία από τις βασικές αρχές της Ένωσης, το υπογραμμίσαμε και σίγουρα δεν μπορεί να υπάρχουν διάφορα μέτρα και σταθμά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βγαίνει στο προσκήνιο οποτεδήποτε υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, γιατί αυτό αποτελεί τμήμα τη προσωπικότητά τη. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εναντί τη Κούβα, απαιτώντα, ζητώντα την απελευθέρωση όλων των κρατούμενων για λόγου συνείδηση στην Κούβα και να υπάρξει σεβασμό των δικαιωμάτων ανθρώπου εκεί. Όχι μόνο αυτό ωστόσο. Πρέπει να δουλέψουμε με αποτελεσματικότητα, να είμαστε αποτελεσματικοί, να πετύχουμε αποτελέσματα που θα βελτιώνουν την ευημερία και τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων, κάτι και επιπλέον την απελευθέρωση. Ε, κάτι μπορούσε να επιτρέψει την απελευθέρωση σε κάποιε περιπτώσει. Μερικέ περιπτώσει όντω υπήρξε πρόοδο. Και υπήρξε πρόοδο διότι ένα βασικό στοιχείο τη πολιτική τη Ένωση εναντί τη Κούβα είναι ο πολιτικό διάλογο με την Κούβα που ξεκίνησε εκ νέου πριν από λίγο, πολύ καλά κατά την άποψή μου έκανε και ξεκίνησε και που επέτρεψε να πάψουν οι κυρώσει που αποτελούσαν τμήμα των θέσεων της Ένωσης και που δεν είχαν κανένα νόημα ο πολιτικός αυτός διάλογος που ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, επέτρεψε να κάνουμε σε λίγο χρόνο κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε από το 2003. Να μιλήσουμε δηλαδή με τις κουβανικές αρχές για τους, πολιτικού για πολιτικούς Και βεβαίως η αξιολόγηση που έκαναν ορισμένοι συναδελφοί σα για το αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού θα πρέπει να γίνεται. Περιοδικά. Θα πρέπει να κάνουμε την ίδια χρονιά αξιολόγηση της διαδικασίας. Πολλοί συνάδελφοί σα, ο κύριο Μάουρο, ο κύριο Γιάννεθ, ο Λουί Μισελ, υπογράμμισαν την σημασία του διαλόγου και τη συνεργασία, αλλά και την ικανότητα και την ηθική, το ηθικό βάρος της Ένωσης για να μπορέσει να τεθεί ως συνομιλητής με την Κούβα και να πετύχει πρόοδο. Γιατί περί αυτού πρόκειται εν τέλει. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την συμφωνία την καταπλειοψηφία συμφωνία που έχει επιτευχθεί στο Κοινοβούλιο σε σχέση με την κατάσταση των δικαιωμάτων των ανθρώπων στην Κούβα, που συνοψίζεται, νομίζω, σε ένα μήνυμα. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο με την Κούβα, ωστόσο η Ένωση θα συνεχίσει να διεκδικεί την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων εκεί και το σεβασμό των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών της Κούβας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και για να τελειώσει η συζήτηση θα δώσω βεβαίω το λόγο στην Επιτροπή στον κύριο Πίλμπακ. Κύριε Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έδειξε ότι αποτελεί λαμπρό αστέρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. πιστεύουμε ότι αν έχει κανείς ισχυρές απόψεις πρέπει να τις καθιστά γνωστές για αυτά τα θέματα. Όπως επίσης γνωρίζετε η βάση τη δουλειά μας με την Κούβα θα παραμείνει η κοινή θέση του 2006 είναι μια στέρεη βάση και να την αλλάξουμε θα πρέπει να σημειωθούν και σημαντικές μεταβολές στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Ο επικοδομητικός διάλογος που ξεκίνησε το 2008 ε, φέρνει αισιόδοξα αποτελέσματα. Δεν έχουμε σημειώσει ουσιαστικές επιτυχίες αλλά σε ορισμένα θέματα σημειώθηκαν πρόοδοι. Και αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να συνεχιστεί. Επίσης και οι επαφές με την κοινωνία των πολιτών. Η Επιτροπή θα ακολουθήσει τα συμπεράσματα του, του Συμβουλίου που λέει ότι θα, οι επαφές με την κοινωνία των πολιτών θα αποτελέσει μέρος επισκέψεων υψηλού επίπεδου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Έχω λάβει 7 προτάσεις ψηφίσματος κηρύσω λοιπόν τη λήξη της συνεδρίασης η οποία θα ξαναρχίσει στις 6 με θέμα της ερωτήσεις προς το Συμβούλιο.